Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Τινησία. Θα επακολουθήσει αυτή αμέσω δήλωση της Επιτροπής και θα μιλήσουν ε, και οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, μην εγκαταλείπετε ακόμη την αίθουσα. Μείνετε δύο λεπτά ακόμα. Mr. Schultz. Κύριε Σούλτς, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μην φεύγετε. Για δύο λεπτά παρακαλώ, μείνετε. Κυρίες και κύριοι, Υπήρξαμε μάρτυρες και με φόβο αλλά και με ελπίδα τα πρόσφατα γεγονότα στην Τινησία. Διοργανώθηκαν ειρηνικέ διαδηλώσει, οι οποίε όμω μετατράπηκαν σε βιε συγκρούσει. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα θλιβερό διότι οι Τινησιακέ αρχέ στράφηκαν κατά των πολιτών τη χώρα. Σήμερα λοιπόν ε, θυμόμαστε, τα θύματα αυτή τη βία αυτών των συγκρούσεων. Εκφράζουμε τη συμπάθεια και τα συλληπιτήριά μα στι οικογένειε των θυμάτων, ιδίω τόσο νεαρών σοβαρών θυμάτων, όπως ε, του Μοχάμετ Μπουαζίζη. Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν, ένα τραγικό συμβάν το οποίο ε, νομίζω σηματοδότησε βαθιά το δημοκρατικό κίνημα στην Τινησία. Ζητήσω λοιπόν να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή και σας παρακαλώ να ηγερθείτε. Thank Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η επιχείρηση του Γιασεμιού. Πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία. Θα ήθελα να σχολιάσω ότι η αποφασιστικότητα και το σθένος του λαού της Τινησίας ε, που ξεκίνησαν αυτό το κίνημα γιατί πρόκειται για την απαρχή βέβαια μιας πολύ μακράς πορείας και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζουμε τους Τινήσιους με κάθε δυνατό τρόπο και από κάθε δυνατή πλευρά θέλουμε να επιτύχουν, θέλουμε να ευτυχήσουν. Εμείς στην Ευρώπη είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία του λόγου ε, και της έκφρασης, τον πραγματικό πλουραλισμό. Θα πρέπει ο λαός της να διαμορφώσει το δικό του μέλλον. Δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι. Θέλουμε όμως και οι αλλαγές να λάβουν χώρα με ειρηνικό τρόπο, να υπάρξει μια ειρηνική μετάβαση να υπάρξει μια κυβέρνηση βασισμένη στο κράτος δικαίου. Απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις αρχές για απελευθέρωση των κρατουμένων, όλων των κρατουμένων. Ζητούμε να διεξαχθεί η σωστή ανεξάρτητη έρευνα σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις διαφθοράς και χρήσης βίας και ζητούμε να γίνουν δίκαιες και ελεύθερες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ε, υπό την παρατήρηση από, διεθνή, από τη διεθνή κοινότητα, από διεθνείς παρατηρητές. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να εκλεγεί μια, ωραία, μια σωστή κυβέρνηση, η οποία θα είναι κυβέρνηση εθνικής ενότητας και θα εκπροσωπεί όλο τον πληθυσμό. Πρόκειται για εταίρους μας, πρόκειται για γείτονές μας. Η εταιρική σχέση θα πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού όχι μόνο του λαού της Τινησίας όμως, αλλά και των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε τους Τινήσιους στο δρόμο για την αλλαγή. Θέλουμε η προσπάθειά τους να στεφθεί με επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, ας στηρίξουμε το λαό της Τινησίας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και τώρα θα διεξαχθεί μια σύντομη συζήτηση ο κύριος Εύτοβιτς, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πάρει τον λόγο σαν πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε και κύριοι βουλευτές, η πρόσφατη λαϊκή εξέγερση στην Ισία είναι άνευ προηγουμένου στην σύγχρονη ιστορία της χώρας. Στις 17 ε, Δεκεμβρίου ένας ε, νέος από αυτό του Πανεπιστημίου αυτοπερπολήθηκε λόγω... από απαλπισία όταν η αστυνομία κατέσχεσε τα φρούτα και λαχανικά που πουλούσε για να ζήσει. Σε λιγότερο από ένα μήνα οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατέληξαν στην αποχώρηση του Προεδρού Μπέναλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την βία και την καταστολή των τελευταίων ημερών του καθεστώτος. Βεβαίω η κατάσταση παραμένει ασταθής. Λαϊλασία και βία ακόμη ξεκολουθούν να αναφέρονται. Η ισία παραμένει σε μία λεπτή φάση, αν και πρώτε ειδήσει για το σχηματισμό κυβέρνηση Εθνική Εθνικής φαίνεται πως φτάνουν σε εμά. Παρά την αβεβαιότητα, το μήνυμα του λαού της Τινησίας είναι σαφές η Τινησία θέλει να είναι μια σταθερή δημοκρατία με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Θέλει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Θέλουν να γράψουν μια νέα σελίδα στην ιστορία τους και θέλουμε να τους υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ο σεβασμός του συντάγματος και τα βήματα τα οποία λαμβάνονται αυτή τη στιγμή για να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα υπενθύμιζε στην Τινησία της διεθνείς της υποχρεώσεις στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Από την αρχή της θητείας μου από την ακρόασή μου ακόμα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανέλαβα πως οπωσδήποτε οι ενισχυμένες σχέσεις σημαίνουν και ενισχυμένες δεσμεύσεις στις σχέσεις μας με την Τινησία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το τόνισα αυτό σε όλες μου τις επαφές με τις αρχές Τινησίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώ πρέπει δηλαδή να έχουν αποτελέσματα όσον αφορά τι δεσμεύσει του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην πρώτη φάση των ε, διαπραγματεύσεων για το καθεστώ ε, τη εταιρική μα σχέση, επέμεινα με τον σαφέστερο τρόπο πω οποιαδήποτε χρήση του άρθρου 61α, του νέου άρθρου 61α του ποινικού κώδικα θα θεωρηθεί από εμάς ασύμβατη με το καθεστώς της εταιρική μας σχέσης και τις κοινέ μας αξίες. Και εάν υπάρχει ακόμα κάποιος και στις δύο πλευρές που θεωρεί πως οι αξίες αυτές ήταν μόνο θεωρητικές, πρέπει να ακούσουν ξανά και ξανά τη φωνή του λαού της θυμησία, τους δρόμους τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Τι ήταν αυτό αν δεν ήταν έτοιμα για δημοκρατία και οικονομική δικαιοσύνη. Όπως είπα εγώ και η κάθε άστον σήμερα το πρωί, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει μια πραγματικά δημοκρατική εκλογική διαδικασία με εγγύηση. Και ελπίζουμε οι λεπτομέρειες να μπορέσουν να ανακοινωθούν το στομότερο δυνατόν μόλις σχηματιστεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε άμεση βοήθεια για να προετοιμάσουμε και να διοργανώσουμε την εκλογική διαδικασία καθώς και διαρκή στήριξη σε μια μετάβαση στη δημοκρατία. Επίσης, εργαζόμαστε σε ένα ευρύτερο πακέτο βοήθειας ε, μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση με, μεταξύ άλλων, οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά προβλήματα της νεολαίας της Τινησίας και εδραίωση του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης και οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη μας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας βασίζεται σε βασικές αξίες που μοιράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους της. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και ανοιχτή οικονομία της αγοράς για να οικοδομήσουμε από κοινού μια κοινή περιοχή, ένα κοινό χώρο δημοκρατίας, σταθερότητας και ευημερίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα τόνιζε πως οι εξής αυτές είναι βασικό τμήμα της πολιτικής γειτονίας μας και προς Νόδο και προς Ανατολάς. Με την ισχυρή μεσαία τάξη της, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την εγκύτητα στην Ευρώπη και τη γενικότερη μετριοπάθειά της, η Τινησία είναι σε καλή θέση για να κάνει το άλμα προς την δημοκρατία το οποίο ζήτησε ο λαός με τόσο σθένος και κουράγιο. Και νομίζω πως όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και συμφέρον για να υπάρχει μια ισχυρή σταθερή δημοκρατική την Έχουμε μακρές και ισχυρές σχέσεις με την Τινησία, μεταξύ των λαών και των επιχειρήσεών μας. είναι η φιλοδοξία της Αντιπροέδρου της ΥΠΑ Εκπροσώπου και να ενισχύσουμε αυτές, να ενισχύσουμε αυτές τις διμερείς σχέσεις με βάση την ορθή διακυβέρνηση, το σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και της κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν έτσι ώστε να γίνουν οι φιλοδοξίες του λαού της νησίας πραγματικότητα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα εκ μέρους του ΕΛΚ Χωσέ Ιχνάσιο Σαλαφράνκα Σάντσες Νέρα. Έχει το λόγο. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Τίνιδα νομίζω ότι μας καλούν να σκεφτούμε πολύ με αίσθημα ευθύνης δύο συγκεκριμένα πτυχές Πρώτα απ' όλα, το κατά πόσον οι πολιτικές στήριξης ε, του status quo ε, σε χώρες οι οποίες δεν προωθούν τις δημοκρατικές αξίες, ε, προωθούν τη σταθερότητα στην περιοχή την ευρύτερη. Και δεύτερον, κατά πόσον κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την εξαφάνιση από την πολιτική σκηνή του κυρίου Μπεναλή. Αρκεί ως προϋπόθεση αυτό για να έχουμε μια πραγματική δημοκρατική μετάβαση στη χώρα. Κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Πρόεδρε, η απάντηση στα δύο ερωτήματα είναι αρνητική. Εξού, ε, κύριε φίλε, θεωρώ ότι πρέπει να προβληματιστούμε ε, και να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε μέσα στο πνεύμα της συνθήκης της Βαρκελόνης να εξηγήσουμε γιατί ο μηχανισμός γειτονίας δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Δεύτερον, όπως μας δείχνει η εμπειρία μας και υπάρχουν ήδη πολλά τέτοια παραδείγματα, όταν υπάρχει κενό εξουσίας οι πιο ριζοσπαστικές και εξτρεμιστικές πολιτικές ομάδες είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά ε, παίρνουν ως όμοιρο την όλη δημοκρατική διαδικασία. Αν θέλουμε λοιπόν να προασπίσουμε τη δημοκρατία ε, πρέπει ε, να αφήσουμε κατά μέρος οποιαδήποτε εξτρεμιστική τάση. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις και προσπάθειες ώστε να μην διολυστήσει αυτή και να μην εξτροχιαστεί αυτή η προσπάθεια. Σωστά είναι όλα αυτά που είπατε. Πρέπει να στηρίξουμε την Ισία και την Τίνο, αλλά θα πρέπει να στείλουμε και μια αποστολή παρατήρηση των εκλογών για τι εκλογέ. Όχι μόνο λόγω τη ηθική επιτακτική ανάγκη που είναι γεγραμμένο, θα έλεγα, στον ίδιο το γενετικό κώδικα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε και εμεί συμφέρον. Αν πηγαίνουμε εμείς στη business, τι νόημα έχει αν στην economy είναι ένας επιβάτης που στις βαλίτσες του έχει μία βόμβα. Εκ μέρους των σοσιαλιστών, ο Πιέρα Αντώνιο Παντσέρη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες για τα τεκτενόμενα στην Τινησία και εκφράζουμε τη θλίψη μας για όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Η νέα φάση είναι συγκεχημένη αυτή που ξεκινάει μετά τη φυγή του πρώην Προέδρου Μπεναλή. Τώρα θα πρέπει να πετευθεί ο στόχος που ζητήθηκε παντού. Οι οικονομικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού και διεύρυνση της δημοκρατίας, των χώρων δημοκρατίας. Πρέπει να, η κοινωνία των πολιτών και αντιπολίτευση ε, να μπορεί να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να διαλέξει το δρόμο της, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε διότι αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και να γίνουν πραγματικές αλλαγές και να μην είναι απλώς εικονικές. Αυτά που συμβαίνουν στην Τινησία αυτές τις μέρες Μα δημιουργούν ερωτηματικά, θέτουν ερωτήματα προ την Ευρώπη και προ εμά για τι καθυστερήσει και τα σφάλματά μα. Το 1995 στη Βαρκελόνη η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το πρόγραμμα τη εταιρική σχέση με τη Μεσόγειο, που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει οικονομική, πολιτική, στατιωτική συνεργασία και κοινωνική και ανθρωπιστική συνεργασία. Αλλά που ούτε ένα από του βασικού στόχου επετεύχθη για την οικονομία. Είχαμε αναδιάθρωση των περιφερειακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων υποδομέ, διότι οι χρηματοδοτήσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν έφτασαν εκεί που έπρεπε και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πόλη είναι στο stand-by. Η υπόσχεση για ζώνη ελευθέρων συναλλαγών δεν υπάρχει. Αλλά η πιο φοφανή χρεοκοπία είναι στο πολιτικό επίπεδο. Αυτού πρέπει να έχουμε επίγνωση, κύριε Επίτροπε. Η Ένωση για τη Μεσόγειο που ξεκίνησε το 2008 παρέμεινε κάτι εικονικό. Η Σύνοδο Κορυφή που θα έπρεπε να διεξαχθεί το Νοέμβριο του 2010 ανεβλήθη επαόριστον. Το πρόβλημα είναι ότι οι διάφορε ευρωπαϊκέ κυβερνήσει δεν βλέπουν συμφέρον για κάποια πραγματική συνεργασία. Θέλουν να κρατήσουν ε, σχέσει με αμφισβητήσιμε ε, κυβερνήσει, εκμεταλλευόμενε τον πλούτο το φυσικό τη χώρα, χωρί ε, δημοκρατία, ενώ οι λαοί ζουν χωρί προοπτική. Και τα προβλήματα ελέγχου τη μετανάστευση είναι όλο και πιο δύσκολα. Δεν θα πρέπει να κλειστόμεθα αν λόγω τη οικονομική και κοινωνική κρίσεω οι διαδηλώσει στην Τινησία μετατράπηκαν σε ένα τσουνάμι που μπόρεσε ε, να πλήξει την εξουσία. Δεν ε, δεν ισχύει πλέον, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο πολιτικός ρεαλισμός της Ευρώπης για αντιμετώπιση του φόβου της ε, Ισλαμικής προσέγγιση. προσέγγισης. Δεν θα πρέπει να ακολουθούμε απεικιοκρατική προσέγγιση από τη σχέση με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ξεκινώντας από τη Βαρκελόνη χρειάζεται ένα νέο όραμα προς τον Νότο, προς τη Μεσόγειο με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό σημαίνει και το ζητώ στεναρά αυτό κύριε Επίτροπε, βαθιά ε, επανεξέταση των πολιτικών εταιρική σχέσεως και γειτονία. Δεν μπορούμε να κρύβουμε το ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο ήταν έτοιμοι να συζητήσουν με την τη συμφωνία για το ε, βελτιωμένο καθεστώς. Ε, και όλα αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν. Χρειάζεται μια αλλαγή γραμμή, χρειάζεται αλλαγή βήματο και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και το λέμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο με μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην υλοποίηση και εφαρμογή μια ιδέα ε, εταιρική σχέση με τι χώρε των νοτίων ακτών τη Μεσογείου. Δεν είναι μόνο προ όφελο αυτών των χωρών, αλλά κυρίω προ όφελο τη Ευρώπη. Πολλά προβλήματα που έχει η Ευρώπη θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν μέσω παραγωγική σχέσεω, σωστή σχέσεω με τι χώρε του Μαγκρέμ. Είναι στενό ο δρόμο, αλλά είναι μοναδικό. Δηλαδή, υποστήριξη οικονομικών και δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, δοθούν όλα τα δύο κατά του φονταμεταλισμού και τη τρομοκρατία. Και ελπίζουμε από, την, από το πικρό μάθημα, το δυνηρό μάθημα τη ε, Ισία, όλα αυτά να είναι χρήσιμα για μα, για να έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση τι είναι χρήσιμο να αλλάξουμε, τι είναι χρήσιμο να κάνουμε και να αλλάξουμε στην δράση την ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ, συνάδελφε για τα σχόλιά σας. Η κυρία Σάκε, για τους φιλελεύθερους, έχει το λόγο. κυρία Σάκε. Ah, Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε, Επίτροπε Φιούλε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ το λαό της για την γενναιότητα και την αντίστασή του όταν τάστε υπέρ των ευκαιριών και της ελευθερίας. Και ελπίζω να μην υπάρχει ελπία και να έχουμε σύντομα δίκαιες εκλογές. Οι πολίτες μίλησαν κατά ενός ε, καταπιστικού καθεστώτος που χρησιμοποιεί σε σφαίρες για να σκοτώσει τους νέους. Μόνο οι αδύναμες κυβερνήσεις το κάνουν αυτό όταν έχουν αποκτήσει διεθαρμένη εξουσία και πλούτο. Τα καθεστώτα λούν να από το να φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών, όχι με το να κλείνουν πανεπιστήμια και την πρόσβαση στην ελεύθερη πληροφόρηση. Με την ε, πρόσβαση στην πληροφόρηση, για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το οποίο γίνεται όλο και πιο σημαντικό για την αντίσταση των λαών στον κόσμο. Εγώ έτσι έμαθα για την εξέγερση αυτή και διάβασα αναφορέ για το τι γίνεται εκεί πέρα και χρειάστηκε ένα ολόκληρο μήνα μέχρι να το αναφέρουν τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το τι γίνεται στον δρόμο. Την ίδια εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, ο Γάλλος υπουργό Εξωτερικών προσέφερε βοήθεια στην Τινησία υπομορφήν ΜΑΤ. Ποια είναι η, αντίσταση, η, η αντίδραση της Κομισιόν σε αυτή την παροχή βοήθειας. Η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του λαού της Τινησίας έλαβε χώρα και στο δρόμο και στο διαδίκτυο η κυβέρνηση της Τινησίας ήταν ε, μία από τις κυβερνήσεις οι οποίες ε, χρησιμοποιούσαν το πιο προχωρημένο software φιλτραρίσματος του διαδικτύου και τον τελευταίο μήνα κατέβαλε κάθε προσπάθεια να καταπιέσει τον κόσμο και μέσω αυτών των τεχνολογιών και βέβαια θα το κάνουν αυτό όλα τα καταπιεστικά καθιστώτα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι η μέρα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ της ΕΠΑ ο οποίος είχε πει φτάνει μια στιγμή κατά την οποία η σιωπή είναι προδοσία. Κύριε Επιτροπέ, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η ΕΠΑ. Έχουν χάσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας τους στον αγώνα για ελευθερία του διαδικτύου. Εμείς έχουμε ακόμα μια μάχη που έρχεται μπροστά μας όταν θα συζητήσουμε τους ε, νόμους της Ουγγαρίας. Αλλά είναι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κοιτούν το συμβολικό παράδειγμα της Τινησίας και θέλουν στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα παίξουμε ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση των ελευθεριών και στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κομμεντή, το πρόεδρος των Πρασίνων. Αγαπητοί συνάδελφοι, ομολογώ ότι θα προτιμούσα το κοινοβούλιο μας ε, να είναι στο ύψος ε, της υπερηφάνειας των τινήσεων ε, που έριξαν τον δικτάτορα Μπεναλή. Έπεσε ο δικτάτορας κυρίες και κύριοι, όμως η δομή της δικτατορίας εξακολουθεί να εφίσταται στην Τινησία. Και σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου εδώ επί χρόνια στήριζε τη δικτατορία και ως δομή και στην Τινησία συγκεκριμένα. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα οι περισσότερες πολιτικές ομάδες αρνούνταν τη διεξαγωγή διαλόγου για την Τινησία αρνούνταν την καταδίκη του Μπεναλή. Αυτό που έκανε η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι παρά το τελευταίο παράδειγμα ε, της συνενοχής της Δύσης. Και για ποιο λόγο λόγω φόβου. Φοβούνταν τον ε, Ισλαμισμό. Όταν είδαμε όμως αυτούς τους ανθρώπους, όταν είδαμε τους τιμήσιους, οι οποίοι δεν ήταν Ισλαμιστές, δεν είχαν κανένα τέτοιο χαρακτηριστικό, αλλά αγωνίζονταν για την ελευθερία τους. Και ο κύριος Μποαζίζη, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε ε, θυσιάστηκε για την Τινησία, ε, τον ακολούθησε όλο το κοινοβούλιο και εμείς ε, δεν δείξαμε την ίδια ικανότητα να σταθούμε πίσω από τον Μπουαζίζη. Να πως έχουν τα πράγματα. Τώρα λοιπόν πρέπει να δράσει η Κομισιόν, να πει ένα πράγμα πολύ απλά, να πει στους Τινήσιους δημοκρατικές εκλογές σε μια χώρα η οποία μόλις εξήλθε από τη δικτατορία δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε δύο μήνε. Δεν υπάρχει βάση, δεν υπάρχουν θεμέλια δημοκρατία, ελευθερία έκφραση, τα μέσα μαζική ενημέρωση, ράδιο, τηλεόραση. Δεν υπάρχουν. Ένα κρατικό τυπογραφείο υπάρχει μόνο. Γι' αυτό ζητάω από την Κομισιό να πάρει τα χρήματα από τη Συμφωνία Σύνδεση και να τα βάλει στην υπηρεσία τη ελευθερία έκφραση τη Τινησία και όχι στην υπηρεσία τη κυβέρνητική οργάνωση τη Τινησία. Δεύτερον, η μεταβατική κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Γιατί, Γιατί η πλειοψηφία αυτών οι οποίοι αγωνίστηκαν ή που είναι εξόριστοι δεν έχουν γυρίσει ακόμη, δεν έχουν αναγνωριστεί. Άρα θα χρειαστεί χρόνος ώστε οι δημοκρατικές δυνάμεις να μην είναι δυνάμεις που είχε αναγνωρίσει εντό αγωγικών ο Μπεναλή, να είναι πραγματικές δημοκρατικές δυνάμεις, να μπορέσουν να αναπτυχθούν πραγματικές δημοκρατικές δυνάμεις στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει ότι για εμάς αυτό τα οποία συμβαίνουν στην την Ισία είναι το κλειδί της κατανόησης και της ελπίδας για όλους τους αραβικούς λαούς. Για όλους τους αραβικούς λαούς. Δημοκρατία και Ισλάμ θα συμβαδίσουν. Μόνο όμως εφόσον εμείς είμαστε ικανοί να στηρίξουμε την ε, δημοκρατία στην Τινησία, η οποία είναι στα σπάργανα και γεννάται αυτή τη στιγμή διότι αλλιώς και, παντού μάλλον θα χρειαστεί να εξεγερθούν, θα πρέπει να εξεγερθούν οι λαοί κατά των δικτατόρων. τι μας δείχνουν οι τινήσεις, δηλαδή ένα μέρος του αραβικού κόσμου, ότι η ελπίδα, η ελευθερία που είδαμε και το 89 ε, στις χώρες Ανατολής, βλέπουμε να γεννάται η ίδια ελπίδα σε μια χώρα όπως η Τινησία, αύριο θα είναι η Αλγερία, μεθαύριο η Αίγυπτος, η Ορδανία. Είναι λοιπόν ε, αδιανόητο για όλους αυτούς τους λόγους να μείνει καθιστό και με σταυρωμένα χέρια το κοινόβιο και να λέει μπορεί ίσως δεν ξέραμε και το 89 τι θα γινόταν με την Πολωνία. Δεν ξέραμε με τον Κορμπατσόφ τι θα γινόταν η Ρωσία. Εάν κάθε φορά που ζητούν οι λαοί ελευθερία τους ζητούμε διασφαλίσεις, τους λέμε να μας πούνε ότι είναι σίγουρο ότι θα πάνε τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξουμε την δημοκρατία. Ποτέ δεν πρόκειται να στηρίξουμε τη δημοκρατία. Εξού και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί. Κουνηθείτε, δείξτε στους τιμήσιους ότι τώρα η Realpolitik είναι η πολιτική στήριξη της δημοκρατίας και όχι πια της δομής της δικτατορίας. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της ομάδας των Πρασίνων εκ μέρους των συντηρητικών ο κ. Σαλ Τάνοκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, η αναταραχή στην Τινησία σίγουρα αντικατοπτρίζει την απογοήτευση και την απελπισία του λαού όσον αφορά την πολιτική και οικονομική αποτρεμά τη χώρα. Η διαφθορά και ο πλούτος τη κυβερνούσα ελίτ ήταν σε πλήρη αντίθεση με τους επίπεδα ανεργία και φτώχεια μεταξύ των απλών ανθρώπων. Ο πρώην πρόεδρο Μπεναλή πλήρωσε το νότο τίμημα διότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στι προσδοκίε ε, των και ελπίδε των λαών του. Του λαού του. Εγώ δεν συμφώνησα με κάποιε εξολογήσει που εξέφρασε πράσινη, εξέφρασαν πράσινοι ότι είναι η πιο καταπιαστική κυβέρνησή του στον αραβικό κόσμο. Η Τινησία ήταν ένα παράδειγμα κατά κάποιο τρόπο μια σύγχρονη κοσμική ε, αραβική χώρα. Η, η πολυγαμία είχε απαγορευτεί. Ε, το τσαντό είχε απαγορευτεί. Είχαν, ο είχε απαγορευτεί κλπ. Λοιπόν, ε, και δεν μπόρεσε να υπονομευθεί κοσμικό, το κοσμικό κράτο. Οπότε οι, ηγέτες της, οι νέοι ηγέτε τη Τινησία που θα βγουν τώρα θα πρέπει να προστατεύσουν αυτή την κληρονομιά και κάποιοι από του ακρεφνεί σίγουρα θα προσπαθήσουν να υποφεληθούν από το χάο και την αναταραχή ε, για να προωθήσουν τα επικίνδυνα προγράμματά τους που προφανώς είναι κάτι που απειλεί την, τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Η νέα πολιτική ηγεσία της Τινησίας θα πρέπει να καταλάβει την κακή διακυβέρνηση και τις τεράστιες ανισότητες που αυτά δημιουργούν βία ριζοσπαστική προσέγγιση στα προβλήματα. Έχουν υποσχεθεί, ε, θα πρέπει να υποσχεθούν μεταρρυθμίσεις διότι μεταρρυθμίσει θα ενισχύσουν τι σχέσει τη Τινησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν μεταξύ, ομάδα μου ζητεί την μέγιστη αυτοσυγκράτηση των δυνάμεων ασφαλεία και τη σύλληψη και δίκαση των τη ηγεσία των προεδρικών φρουρών του παλιού καθεστώτο που ήταν υπεύθυνοι για του πρόσφατου πυροβολισμού που πυροβόλησαν αθώου ε, πολίτε σε μια μάταιη προσπάθεια να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και συγχαίρω τον επαγγελματισμό του στρατού που προστάτευσε ε, του θεσμού τη δημοκρατία. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσουμε στη νέα την ισιακή κυβέρνηση ενότητα κάθε βοήθεια και επίση να δώσουμε κάθε βοήθεια στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως που απομονώθηκαν εκεί ε, λόγω του ότι είχαν πάει εκεί για διακοπές. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς. Η Μαρή Κριστίν Βερζόν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με κάποια υπερηφάνεια και μεγάλη συγκίνηση μιλώ σήμερα σε αυτό το κοινοβούλιο εν ονόματι της ομάδας μου της Ευρωπαϊκής Συνοτικής Αριστεράς και θα ήθελα να πω ότι ήμασταν λίγοι και λίγες θα έλεγα που, που καταγγείλαμε την παρέκκληση του καθεστώτος της νησίας και αυτά που έκανε σε εκείνους και εκείνες που τολμούσαν να επικρίνουν την κυβέρνηση και να καταγγείλουν τι πρακτικέ που ακολουθούσε και κυρίω τα βασανιστήρια των προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έπρεπε ένα νέο 26 ετών να καταναλωθεί από τη φωτιά για να εξεγερθεί ο λαό τη Τινησία, να, μην να μην φοβάται πλέον, διότι αισθανόταν μόνοι του. Το πνεύμα τη ελευθερία γεννήθηκε. Έπρεπε να περιμένουν πάνω από 50 νεκρού να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που ζήτησε την αυτοσυγκράτηση εκείνων που χρησιμοποιούν τη βία χωρίς να αμφισβητεί την ε, ακαθαγιασμένη εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την Ισία και χωρίς καταδικάζει τη βία παρά μόνο μετά το Σάββατο. Και το λιγότερο που πρέπει να πούμε είναι ότι το καθεστώς της Τινησίας δεν σας άκουσε από όταν είχατε ε, διοριστεί. Αυτό το μήνυμα για την αυτοσυγκράτηση ε, μου κάθεται στο λαιμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σιωπηλό ε, μια μετριοπαθή ανακοίνωση στην ε, ομάδα του Μαγκρέμπ έκανε. Μόλις, τα, μόλις το Σάββατο μίλησατε κύριε Πρόεδρε και σήμερα η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρνήθηκε ένα γραπτό ψήφισμα. Οι ευρωπαϊκές αρχές γνωρίζουν ε, να είναι πιο οξύς ε, έναντι άλλων καθεστώτων. Ξέρω ως Γαλλίδα ποιες είναι οι ευθύνες της γαλλικής κυβερνήσεως και δεν θα αναφερθώ ξανά στα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών μας ε, προφανώς για κάποιους η ώρα των απικιών δεν έχει φύγει πια αλλά ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι του παρελθόντος. Χάρη στο θάρρος του τινησιακού λαού σε μερικές ημέρες το τινησιακό θαύμα ε, κατέρευσε και έδειξε την πραγματική του όψη. Αυτό που αγαπούσαν πολύ εδώ. Σήμερα ε, είναι μεγάλη τεράστια ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πρέπει άνευ αναμίξεως να συνοδεύσει τον τυνησιακό λαό στη μετάβασή του στη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθήσει τις εκλογικές διαδικασίες, να φροντίσει ούτως ώστε μια επιτροπή έρευνας ανεξάρτητη να ρίξει φως σε όλα όσα συνέβησαν ε, στις βιοπραγίες, στη διαφθορά ο λαός της Τινησίας δεν θα πρέπει πλέον να αποτελεί αντικείμενο λαφυραγώγησης από οικογένειες όπως τον Μπέναλή θα πρέπει τα αγαθά του Μπεν Αλή να ε, κατασχεθούν. Θα πρέπει τελικά να αποκτήσουν σιγά σιγά εμπιστοσύνη την ίση. Ε, δύσκολα είναι τα πράγματα ακόμα σήμερα και μπορεί να ε, βγουν παραδείγματα για το Μαγκρέμπ από αυτά που συμβαίνουν στην Τινησία. Ξέρουμε παρόμοιε εξαγέρσει μπορούν να γίνουν σε όλε αυτέ τι χώρε όπου οι δυτικοί πάντα προστατεύουν τα δικά του συμφέροντα και τα θέτουν πάνω από τα συμφέροντα των λαών. Έχουν αυτοπερθεί άνθρωποι και στην Αίγυπτο και στην Αλγερία και στη Μαυριτανία. Θα πρέπει από τι ομιλίε να περάσουμε στι πράξει όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι και η ώρα να αναδιαφθρωθεί η εταιρική σχέση τη Ευρωπαϊκή Ενώση με τι χώρε του Νότου και να υπάρχουν δημοκρατικέ απαιτήσει για τη σύνευση των συμφωνιών. Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητα. Διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τελικά θα παίξει το παιχνίδι των ε, ακρεφνών ισταμιστών. Η ελευθερία και δικατία, ο συνάδελφος κύριος Μπάτεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούζακ, αναφέρατε στην αρχή κάποια πράγματα για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση και ζητήσατε να στηρίξουμε το λαό της την Ισία. Κανένας δημοκράτη δεν διαφωνεί. Οι άνθρωποι ανέχονται πολλά από ανίκανες και διεφθαρμένε κυβερνήσεις, αλλά εάν του πρόξουμε στα όρια θα επαναστατήσουν. Είναι δόγμα των υπηρεσιών εσωτερική ασφαλείας πως οποιοδήποτε πληθυσμό απέχει μόνο τρει μέρες από ταραχές και κοινωνικές αναταρχές όταν τελειώσουν τα τρόφιμα. Μπορούμε να κάνουμε παραλληλισμού μεταξύ Ισίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ανίκανη και μη δημοκρατική κυβέρνηση έχει μια πολιτική τάξη που είναι αποκομμένη από τις επιθυμίες του λαού τη. Υπάρχει υψηλή ανεργία των νέων σε πολλές χώρες στην Ένωση ως άμεσο αποτέλεσμα των πολιτικών της Ένωσης. Υπάρχουν ήδη τάραχες στην Ελλάδα λόγω της ιδεολογικής της προσήλωσης στο ενιαίο νόμισμα. Χώρες όπως η Ισπανία, Πορτογαλία και η Ιρλανδία μπορεί σύντομα να ακολουθήσουν την Ελλάδα καθώς δεν μπορούν να αντέξουν οι οικονομίες τους τον ζουρλομανδία του ευρώ. Μην νομίζετε πως δεν μπορεί να συμβεί στην Ευρώπη. Όταν οι κυβερνήσεις γίνονται εχθρός του λαού τους, ο λαός θα επαναστατήσει. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε στην εισαγωγή σας, κύριε Πρόεδρε, αλλά ας δούμε αυτές τις αρχές να εφαρμόζονται και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφοι των πολιτικών ομάδων που λάβατε τον λόγο και για τα σχόλιά σας και ευχαριστώ και τον Επίτροπο τον κύριο Φιούλε για τα σχόλιά του εξ ονόματος της Επιτροπής.